Έχω την τιμή να πω ότι μόλις αποφάσισε η διάσκεψη των Προέδρων Πολιτικών Ομάδων να δώσει το βραβείο Ζαχάροφ για το 2017 για την ελευθερία της σκέψης στην δημοκρατική αντιπολίτευση της Βενεζουέλα. All'Assemblea Nazionale rappresentata